Βλέπω ότι είναι δύσκολο το πρωινό για όλους. Ας ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία για το κανονισμό για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες ε, για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρέπο. Αντικαθίσταται. να πω δύο λόγια. για κάτι που είναι αρκετά σημαντικό. Πρόκειται για μια τροποποίηση του κανονισμού. Ο χθεσινός τρίμερης διάλογος ε, πήγε πολύ καλά, είχε κάποιο αποτέλεσμα και περάσαμε όλα όσο επιθυμούσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Κομισιόν για την καλή συνεργασία και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για την υποστήριξή τους. Η ιδέα του Κοινοβουλίου ήταν να συμπεριλάβουμε στην πρόταση της Κομισιόν μια ρήτρα αναθεώρησης, μια ρήτρα επαναξιολόγησης, δηλαδή ότι θα έχουμε μια έκθεση για την δραστηριότητα της προστασίας των καταναλωτών μέχρι το 2014. Ο στόχος είναι να δούμε αν ο κανονισμός είναι αποτελεσματικός, να δούμε το μηχανισμό λειτουργίας και ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογή. Και ο στόχος, ε, αν χρειαστεί, είναι να προτείνει η Κομισιόν νέα νομοθεσία πριν από το 2014 το Συμβούλιο όπως και η Κομισιόν ήταν αντίθετη στη συμπερίληψη αυτής της ρήτρης αναθεώρησης, αλλά εν τέλει υποχώρησαν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να περάσει αυτή την νομοθεσία στην πρώτη ανάγνωση. Αν όλα πάνε ως ε, έχουν προβλεφθεί στις 5 Ιουλίου θα έχουμε τη συζήτηση στην Ολομέλεια και στις 6 Ιουλίου θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Μάλιστα, ευχαριστώ. Αν η Κομισιόν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Μολνάρ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ρέπο. Να ευχαριστήσω όλους όλα τα μέλη της Επιτροπής και όλους όσους ε, συμμετείχαν ε, στην συζήτηση για την επιμονή του στο να βρούμε μια λύση και πράγματι μπορώ να επιβεβαιώσω πως η Κομισιόν ε, ε, συμφωνεί με το χθεσινό κείμενο και ελπίζω σήμερα η ψηφοφορία να κυλήσει ομαλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχουμε μια ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ρέπο. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Τώρα, ας περάσουμε στη ψηφοφορία του θέματος τεχνικές απαιτήσει ε, για ε, τις μεταφορές πιστώσεων και των άμεσων χρήσεων σε ευρώ της κυρίας Γκέπαρτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως έχουμε απλή ψηφοφορία και εδώ. Είχαμε πολύ ευχάριστο κλίμα με τους κοιόδης Μια στιγμή να ετοιμαστεί και το ΕΛΚ. Οπότε, ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές Είχαμε πολύ επικοδομητική συνεργασία. Συμφωνήσαμε σε όλα τα ουσιαστικά σημεία. Και συνοψίζοντας, λέμε πως είναι λογικό και για άμεσες ε, χρεώσεις ε, και εμβάσματα να έχουμε μία κοινή προθεσμία για να μην έχουμε διαφορετικές ημερομηνίε στα κράτη-μέλη και είπαμε πως θα πρέπει να δώσουμε 24 μήνες χρόνο στα κράτη-μέλη για την εισαγωγή του συστήματος για να είναι αποτελεσματικό. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα από τον οποίο συμφωνήσαμε. Δεύτερο σημείο συμφωνίας απαιτήσει πληροφόρησης των καταναλωτών και είναι υποχρέωση και των κρατών μελών και των τραπεζών να ενημερώσουν τους πελάτες τους για το τι σημαίνει IBAN και BIC. Από το τι αποτελείται και για το ότι δεν είναι τίποτα το φοβερά δύσκολο. Γιατί ε, αν και φαίνεται πολύ έτσι, μεγάλος αριθμός, Ε, αποτελείται από διάφορα άλλα στοιχεία και δεν είναι τόσο δύσκολο. Οπότε νομίζω μπορούν να βοηθήσει τους ε, καταναλωτές. Επίσης, εάν ε, πάει κάτι λάθος και πρέπει να ξαναμπούν λεφτά στο λογαριασμό, τότε θα πρέπει να πληρώνει μόνο για λάθη για τα οποία είναι ο ίδιος υπεύθυνος ο πελάτης. Για τα υπόλοιπα πρέπει να τα βρουν οι τράπεζες. Νομίζω λογικό είναι να μην επιβαρύνεται ο πελάτης για λάθη μεταξύ των τραπεζών. Νομίζω πως είπατε ουσιαστικά. Επί των οποίων συμφωνήσαμε. Το θέμα να γίνουν τα πράγματα απλά για τους πολίτες. Να δώσουμε στο δυνατόν περισσότερες ε, πληροφορίες για να καταλάβουν το σύστημα ΣΕΠΑ οι πολίτες. Και όπως σας είπα θα δώσουμε άλλα δύο χρόνια για να το εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία και ευχαριστώ τους συναδέλφους και τη γραμματεία. Ε, Οι συγκεκριμένες συζητητές θέλουν το λόγο. Κύριος Μπουζουτήλ καταρχήν. Uh, Πρόεδρε, Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Κέπχαρτ για την πολύ καλή συνεργασία, αλλά θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να κάνω μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία 15. Θα φτάσουμε σε μετέπειτα στάδιο, αλλά ήθελα να το αναφέρω τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν δεν ε, υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Όλοι έχουν ε, την κάρτα. Μάλιστα. Ας κάνουμε τον πρώτο έλεγχο, αν μπορούμε να ψηφίσουμε. Για το ΕΛΚ. Μάλιστα, κλείνει η ψηφοφορία. Σοσιαλιστές. Perfetto. Eh, il gruppo dell'Alde. Φιλελεύθεροι. Perfetto. Io direi che siamo, possiamo... Πολύ ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, πιστεύω. Λοιπόν, τροπολογία 6 της κυρίας Γκέιπαρτ, υπέρ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Ναι, ναι, θα πάμε πιο γρήγορα σε λίγο. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας περάσουμε στο ε, συμβασμό 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν τροπολογία 52 υπέρ άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 15-15. Τροπολογία 48 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ας περάσουμε στην τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία του κ. Μπουζουτήλη, παρακαλώ. Ναι, ναι. από το ΕΛΚ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω αυτή η παραγραφός να μετακινηθεί από το άρθρο 6 στα εκτιμώντας. Δηλαδή, αν το μετακινήσετε στα εκτιμώντας, μπορεί το ΕΛΚ να ψηφίσει υπέρ. Υπάρχουν σχόλια? Δεκτό. Πολύ ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 55 τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε την τροπολογία 57. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται για μία ψήφο. Non avete ancora Δεν ψηφίσατε ακόμα, ας ξαναψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 59. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Ωραία. Απορρίπτεται. 19 κατά. Τροπολογία 60. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 63 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Όχι. Έχουμε. Με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 1 για τα εκτιμώντας. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 1 για τα εκτιμώντας, κύριε Γκέπαρτ. Περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός περιθμών 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν έχουμε τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται 17-17. Τροπολογία 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έχουμε την τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κατόπιν. Έχουμε προφορική τροπολογία της κυρίας Γκέπαρτ αλλά ήδη το βλέπετε στην, στο έγγραφο. Έτσι λοιπόν, αν, θέλετε το, αν δεν θέλετε το λόγο, να συνεχίσουμε γιατί βλέπουμε την τροπολογία στο κείμενο. Να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχουμε μία ακόμα ψήφο από το ΕΣΥΑΡ. Στην αρχή είχαμε τρει. Πέρα στις Απορρίπτεται. Περνάμε στο παράρτημα. Λοιπόν, ε, να ψηφίσουμε την τροπολογία 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Μάλιστα, πέρας, απορρίπτεται. Τώρα, περνάμε στη ψηφοφορία για το παράρτημα. Τροπολογία 31. Περ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, έχουμε την τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Υπέρ 34, μόνο μία αποχή. Συγχαρητήρια, κυρία Γκέπαρτ.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 Παρακαλώ να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θέλω να σας ανακοινώσω μια πρόταση σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία για την οδηγία για τους καταναλωτές. Η πρόταση είναι η εξή. να ψηφίσουμε αύριο το πρωί στι 10 θα έχουμε μία και μόνη ψηφοφορία, πολύ σύντομα δηλαδή. Αντίθετα, σήμερα στι 3 θα έχουμε μία συνάντηση και κλεισμένων των θυρών με του σκιώδη. Θα ήθελα τη δική σας αντίδραση απέναντι σε αυτή την πρόταση, αν συμφωνείτε, αν θέλετε να διατηρηθεί η ψηφοφορία σήμερα στις 3. Παρακαλώ, κύριε Γκέπαρτ. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε ακόμα κείμενα από την Κορεπέρ. Τώρα ακόμα ε, διαβουλεύονται, οπότε δεν μπορούμε να αποφασίσουμε πώς θα ψηφίσουμε. Καλό είναι νομίζω και οι υπόλοιποι βουλευτές ε, να διαβάσουν το κείμενο. Οπότε δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα στις 3. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε στη σημερινή διατύπωση. Possibly vote μωρό Πιθανώς να ψηφίσουμε αύριο. Και αν το κείμενο είναι διαφορετικό από αυτό που συμφωνήσαμε, οπωσδήποτε δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Γι' αυτό η πρότασή μου είναι πιθανώς αύριο στις 10 η ώρα. Μάλιστα, βεβαίως. Ήθελα να συμφωνήσω με την πρόταση αυτή επί της διαδικασίας. Ε, ευχαριστώ και εγώ και εγώ συμφωνώ με αυτή την ε, πρόταση. Να ψηφίσουμε αύριο το πρωί στις 10. Να δούμε τι γίνεται με τα διαπραγματεύσεις πρώτα. Άλλος κανεί. Μάλιστα, κύριε Χαλμπρού. Um, ναι, νομίζω πως ε, λογικό είναι αυτό το οποίο προτείνεται, αλλά έχουμε μισή ώρα το απόγευμα που προτείνω να συνεδριάσουμε και κλεισμένων των θυρών. Μπορεί να έρθει ο καθένας, αλλά βεβαίως ε, κυρίως οι σκιώδεις συγητές, για να έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε το κείμενο και νομίζω πως η Επιτροπή μετά θα αποφασίσει το απόγευμα για το εάν θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί στις 10. Επίσης να τονίσω πως ε, το πρόγραμμα αυτό έγινε έτσι επειδή η διάσκεψη των Προέδρων μας πρότεινε η τελική ψηφοφορία ε, να γίνει στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να μην τηρήσει την συνηθισμένη περίοδο αναμονής. Η δική τους πρόταση είναι αυτή, όχι η δική μου. Α, μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του βεβαίω. απλά θέλω να ξεκαθαρίσω πως η αρχική μας ιδέα ήταν να πάει συνεδρία του Ιουλίου. Εν πάση περιπτώσει αυτό πρότεινε η διάσκεψη των Προέδρων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση της μισής ώρας, αλλά ελπίζω να συναντηθούν οι σκιώδεις ε, πριν από τη συζήτηση αυτή. Και βεβαίω ε, θα το πούμε και τρεις η ώρα με διερμηνία. Ευχαριστώ Γκέπ. Ναι. Συγγνώμη. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία στις 10.30 γιατί έχω και ένα ραντεβού που δεν μπορώ να αναβάλω στις 10. 10.30 αν συμφωνούν και οι άλλοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. 10.30 είναι εντάξει για αύριο. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μία κρόση για αύριο. Θα έχουμε πολλούς ομιλητές δηλαδή. Έτσι νομίζω ότι θα ήταν προβληματικό να ψηφίσουμε στα 10.30. Θα έρθει και ο Υπουργό εδώ από τις 9 ως τις 10 και η δική μου πρόταση ήταν να ψηφίσουμε στις 10 και να ξεκινήσει μετά η ακρόαση. Αν είναι στις 10.30 θα πρέπει να διακόψουμε την ακρόαση για την ψηφορία. Νομίζω ότι δεν είναι και πολύ θετικό κάτι τέτοιο. Κύριε Γκέπερτ, μήπως ε, μπορείτε για μισή ώρα να κάνετε αυτήν την υποχώρηση, να αλλάξετε το πρόγραμμά σας διαφορετικό, διαφορετικά θα διακόψουμε την ακρόαση και νομίζω ότι το οφείλουμε στον ε, κύριο Σλουβίνη και τους υπολείπους να ξεκινήσουμε την ακρόαση εγκαίρως. Κοιτάξτε, δεν είχα δει το πρόγραμμα. Ίσως ε, να ψηφίσουμε λίγο πριν τις 10. Είναι πάρα πολύ γρήγορη αυτή η ψηφοφορία. Γιατί ε, καθώς έχουμε την ακρόαση δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα. Δηλαδή στις 9 αν προτιμάτε. Äh, um äh, um ε, τότε 9, 9 και 4. 9 και 4 είναι καλά. I'm sorry, but uh, it's not... Συγγνώμη. Ε, δεν μπορώ εγώ στις 9. Ε, εγώ χρειάζομαι 10 άμα είναι αύριο. 10 η ώρα. Σε Λοιπόν, ε, θέλετε να ψηφίσουμε για αυτό το σημείο. Πρόεδρε, αν ε, κατάλαβα καλά, νομίζω ότι 5-10 λεπτά θα χρειαστούμε για την ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν θα ήταν δυνατό. Δηλαδή, μέσα σε 5 λεπτά να λύσουμε το θέμα. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. 10 η ώρα, αφού δεν γίνεται αλλιώ. Ε, να δω τι θα κάνω, εν πάση περιπτώσει. Όχι, όχι στις 10. <laughs> Ευχαριστώ την κυρία Γκέμπερ για την ε, διαθεσιμότητά τη. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν ψηφοφορία αύριο που θα είναι πάρα πολύ σύντομη στι 10 αύριο το πρωί. Και επομένω επιβεβαιώνουμε και τη συνάντηση με του σκιώδει συγγητέ σήμερα στι 3. Εντάξει, συμφωνείτε όλοι. Πολύ ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε με την παρουσίαση της μελέτης ε, για ε, την ψηφιακή εσωτερική αγορά για τις ηλεκτρονικές ε, συμβάσεις και τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ροζενκέτερ και στην κυρία Χόφμαν. Ähm, Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Χαιρόμαστε που μπορούμε σήμερα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ε, μελέτης μας. Εγώ είμαι η Γιανέτε Ρόζαν Κότερ και δίπλα μου είναι και η κυρία Χόφμαν. Ανήκουμε στο δικηγορικό γραφείο FPS ε, με τη βοήθεια της κυρίας Γκιούλα Σμιτ από τη Βουδαπέστη ε, συντάξαμε αυτή την έκθεση το γραφείο μας ειδικεύεται στους ε, τομείς ε, της ε, πληροφορικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας και δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της Γερμανίας. Είδαμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ηλεκτρονικές υπογραφές στο πλαίσιο μιας ψηφιακής εσωτερικής αγοράς. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν στα πράγματα τα οποία μας είπατε. Πρώτα απ' όλα δηλαδή το ερώτημα της επεξεργασίας των κανονισμών περί ηλεκτρονικών σημάτων, για τα οποία μιλήσει η κυρία Χόφμαν. Το δεύτερο αφορά την κατάσταση, ε, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή για τις ε, τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις ε, προμήθειες. Οπότε πρώτα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Χόφμαν για την ηλεκτρονική υπογραφή και μετά θα μιλήσω εγώ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι.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 There are three levels of electronic signatures. The simplest form is the simple electronic signature. Ε, το... Η πρώτη ηλεκτρονική υπογραφή που θα εξετάσουμε είναι παραδείγματο η πιο απλή, δηλαδή το όνομά μας ε, μετά από ένα email. Κατόπιν υπάρχει η προχωρημένη ηλεκτρονική, ε, προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ε, χάρη στην οποία μπορεί να πιστοποιηθεί ο υπογράφων και κατοχυρώνεται έτσι η ακαιρεότητα, η γνησιότητα αν θέλετε ενός εγγράφου διότι συνδέεται τόσο άρρηκτα με τα δεδομένα ώστε ε, είναι ανοιχνεύσιμη η αδίποτε αλλαγή γίνει στα δεδομένα μέσα στο έγγραφο. Κατόπιν ναι, η ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, Qualified Electronic Signature, ε, εστιάζεται η οδηγία σε αυτήν την σε αυτού του είδους την υπογραφή πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτήσει της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και επιπροσθέτως θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ειδικό πιστοποιητικό και να έχει δημιουργηθεί με μια ασφαλή συσκευή δημιουργία ηλεκτρονικών υπογραφών. Μπορείτε μέσα στη μελέτη μας να δείτε και άλλες τεχνικές ε, λεπτομέρειες και προδιαγραφές για τις υπογραφές. Υπάρχει σαφέ νομικό καθεστώ που διέπει τις ηλεκτρονικές υπογραφέ θεωρούνται ως τεκμήριο επιστοποίηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Σε σχέση τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις έχουμε την οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή από το 1999 που προσδιορίσε το νομικό πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών και των υπηρεσιών πιστοποίηση. Επίση υπάρχουμε Υπάρχουν ε, πολλοί άριθμα πρότυπα, τεχνικά πρότυπα για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και η βασική δομή για τις ε, ε, λογιστική δομή για τις ηλεκτρονικές υπογραφές με βασικές πληροφορίες για αυτούς που εκδίδουν τα πιστοποιητικά αυτά και το ίδιο σύστημα διέπει και την επιτήρηση αυτών. Currently, electronic ε, οι ηλεκτρονικές υπογραφές χρησιμοποιούνται στον τραπεζικό τομέα, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά δεν χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως ακόμη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχουμε και την Αστριακή ηλεκτρονική κάρτα που ε, ονομάζεται Burger χάρη στην οποία μπορεί ένας πολίτης να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική υπογραφή, ε, ούτω ώστε να ε, χρησιμοποιήσει το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της κυβέρνησης. Παραδείγματος χάρη, επιγραμμικά μπορεί να υποβληθεί ένα αίτημα για συνταξιοδότηση, για παροχές, για έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως και ούτω καθεξής. Στην Εστονία η πλειοψηφία των πολιτών χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές υπογραφές και κινητές υπογραφές ε, κυρίως ε, για ε, τον ηλεκτρονικό τραπεζικό τομέα, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία κτλ. Ε, όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυτή την οδηγία, υφίστανται όμως ακόμη διάφοροι φραγμοί που παρεμποδίζουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών. Ε, μεγάλη ποικιλομορφία υπάρχει από κράτος σε κράτος και γι' αυτό έχουν ε, αναπτυχθεί διάφορες επιμέρους εφαρμογές ε, για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, το οποίο όμως έχει οδηγήσει σε κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς ε, και απώλεια της αξιοπιστίας ηλεκτρονικής υπογραφής, ακριβώς επειδή δεν είναι δυνατή η διασυνοριακή τους χρήση λόγω της έλλειψης διαλειτουργικότητας. Υφίστανται λοιπόν εμπόδιο, μπορούμε να ταξινομήσουμε σε τέσσερις κατηγορίες. Um, barriers at the legal level σε τεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο εμπιστοσύνη και τα πρακτικά ζητήματα, Α δούμε μία-μία τις κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα νομικά ζητήματα. Ε, ποια είναι τα προβλήματα στο νομικό τομέα. Υπάρχουν διαφορές ως προς την εφαρμογή και την ερμηνεία της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Φερρυπίν, ο υπογράφων ορίζεται ως άτομο. Ε, είναι ασαφής ορισμός και άρα δεν ξέρουμε αν μόνο φυσικά πρόσωπα δικαιούνται τέτοια πιστοποιητικά. Αυτό είναι που ισχύει στα περισσότερα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με το αν νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν ηλεκτρονικές υπογραφές στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ουγγαρία, στη Λετωνία και στη Ρουμανία υπάρχει ήδη αυτό ε, στο ένομο σύστημα. Κατόπιν, ε, σύστημα επιτήρησης η οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να κατοχυρώσουν ένα επαρκέ σύστημα επιτήρησης των παρόχων των πιστοποιητικών ε, γνησιότητα. Αλλά επαφείται αυτό στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μέλων και ω εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί διάφορα εθνικά συστήματα και το σύστημα βεβαίω αμοιβαία αναγνώριση κατόπιν ε, με την οδηγία εστιάζουμε στις ε, ειδικέ ηλεκτρονικές υπογραφές και στην έκδοση των ειδικών πιστοποιητικών. Αλλά δεν ρυθμίζεται σαφώς ε, οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χορήγησης πιστοποιητικού ε, που όμως υπάρχει στην αγορά, Παραδείγματο χάρη συμπληρωματικές υπογραφές, ancillary signatures ή οποιασδήποτε πολιτικές σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο εμπόριο και άρα ε, διάφορες υπηρεσίες ε, παραδείγματος χάρη ε, συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες σχετικές με τις ηλεκτρονικές υπογραφές υπηρεσίες δεν καλύπτονται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ηλεκτρονική υπογραφή σε όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πέρα από αυτούς τους φραγμούς σε νομικό επίπεδο, Υπάρχουν άλλα τεχνικά προβλήματα και προβλήματα εμπιστοσύνη. Επίση, ε, μπορώ να πω εδώ ότι υπάρχουν πολλά πρότυπα για τι ηλεκτρονικέ υπογραφέ, αλλά είναι πολύ σύνθετα και ε, δύσχριστα τα, τα συστήματα, δεν υπάρχει σαφής προσανατολισμός, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές και δεν είναι πλήρη τα πρότυπα. Επίσης δεν υπάρχουν προδιαγραφές ε, για να καλυφθούν όλων των ειδών ηλεκτρονικές υπογραφές. Επίσης, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με ηλεκτρονικές υπογραφές από άλλα κράτη-μέλη στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στην πράξη. Εξάλλου υπάρχει μεγάλη δυσπιστία ως προς τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών, ε, διότι δεν γίνονται ευρέως αποδεκτές οι υπογραφές από όλους τους συμβασίουχους, δεν έχουν όλη την απαραίτητη υποδομή για να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπογραφή. Το κόστος της ηλεκτρονικής υπογραφής είναι υψηλό ή δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με το όφελός του και εξακολουθεί ε, να λείπει η απλή εφαρμογή για την χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής που θα προσέλκυε ένα ευρύτερο κοινό. Άρα πρέπει να αναλάβουμε δράση για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και τώρα αντιμετωπίζουμε το εξή θέμα. Η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών πώς μπορεί να αναβαθμιστεί και πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη διασυνορία και τους χρήση. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο έχουν προταθεί δύο βασικά στρατηγικέ από διαφορετικέ μελέτε που ζήτησε να διεξαχθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη είναι η προσέγγιση ευρεία κλίμακα με στόχο τη δημιουργία ενό πλαισίου, νομικού πλαισίου, τεχνικού πλαισίου και πλαισίου εμπιστοσύνη, που θα διέπει τι ηλεκτρονικέ υπογραφέ, επίση τουλάχιστον τη αναθεώρηση ή ενίσχυση τουλάχιστον της οδηγίας ηλεκτρονικών υπογραφών. Η δεύτερη τη οδηγια είναι η προσέγγιση μικρής κλίμακος ε, οι θεασότητες αυτής της προσέγγισης προτιμούν να βελτιώσουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δίχως τροποποίηση δηλαδή της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Η βασική διαφορά των δύο προσεγγίσεων τοποθετείται στο νομικό επίπεδο. Ε, οι οπαδοί της πρώτης προσέγγισης, ευρύω κλίμακος, ε, ε, θα ήθελαν να αναθεωρηθεί αρδίνη η οδηγία περί ηλεκτρονικών υπογραφών, ούτως ώστε να εφαρμόζεται όχι μόνο στις προηγμένε και ειδικέ ηλεκτρονικές υπογραφές και τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως ισχύει τώρα δηλαδή, αλλά να ρυθμίζει όλων των ειδών τις ηλεκτρονικές υπογραφές και σχετικά προϊόντα και όλα τα, όλες τις υπηρεσίες καθώς και τις επικουρικές ως προς τις ηλεκτρονικές υπογραφές υπηρεσίες, καθώς και επιστοποίηση και αναγνώριση. Ε, τώρα για τη δεύτερη προσέγγιση μικρή κλίμακο. Οι οπαδοί τη ε, αντιτάσσονται στην αναθεώρηση τη οδηγία ε, διότι θεωρούν ότι θα είναι μακρά και επαχθή η διαδικασία και ένα άλλο κίνδυνο που ελοχεύει είναι να διαταραχθεί η εύρημη λειτουργία τη αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ένα εγγραφό σχετικά με μια κοινή ομοιόμορφη ερμηνεία τη οδηγία περί ηλεκτρονικών υπογραφών και διευκρινίζει ειδικά ζητήματα. Η οπαδοί και των δύο προσεγγίσεων ε, είναι υπέρ της δημιουργίας ενός, ε, ε, μιας δέσμης προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και θεωρούν ότι οι λεπτομέρειες δεν πρέπει να ρυθμίζονται μέσα στην οδηγία τόσο ώστε να παραμείνει τεχνικώ ευέλικτη αυτή, αλλά ε, προτείνουν μια καταγραφή ε, των νομικών προτύπων μέσα από αποφάσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως συμβαίνει και τώρα. Ε, και τη νομική βάση για κάτι τέτοιο βρίσκεται στο άρθρο 3.5 τη οδηγία. Σχετικά με την εμπιστοσύνη, οι οπαδοί της πρώτης κατηγορίας ε, θεωρούν ε, ότι θα έπρεπε να υπάρχει επιτήρηση και ε, θελούσια πιστοποίηση όλων όσων προσφέρουν οι υπηρεσίε επιστοποίηση. Άρα πρέπει να τίθεται και ζήτημα αστική ευθύνη καθώ και πιστοποίηση για όλε τι υπηρεσίε και δημοσίευση του καταλόγου, ούτω ώστε να υπάρχουν βασικέ πληροφορίε στη διάθεση όλων των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ε, κατόπιν ε, χρειάζονται ε, μέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών υπογραφών βάσει και των δύο θεωριών, της ευρείας δηλαδή και της στενής κλίμακας. Τώρα, Θεωρούμε ότι η προσέγγιση ευρείας κλίμακος ε, είναι η προσφορότερη γιατί θα προσφέρει μια υγιή νομική βάση που θα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπογραφών και άρα πρέπει να γίνει αναθεώρηση της οδηγίας και επέκταση αυτής ε, του πεδίου εφαρμογή της. Θεωρούμε επίσης ε, ότι ένα εξορθολογισμένο νομικό πλαίσιο με ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές είναι μια διαδικασία που έχει ήδη αρχίσει γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει αναθέσει εντολή πιστοποίηση τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης, ε, τυποποίησης, ε, συγγνώμη, και πρέπει να οθεί συνέχεια λοιπόν σε αυτή την εντολή που είναι γνωστή ως M460. Κατόπιν τα πρότυπα και προδιαγραφέ θα καταχωρούνται σε αποφάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι θα πληρούνται και τεχνικέ προποθέσει τη οδηγία. Προτείνουμε επέκταση του άρθρου 3.5 τη οδηγία και εισαγωγή επιπροσθέτων απαιτήσεων σχετικά με τη νομική συμμόρφωση ω προ τα προϊόντα και υπηρεσίε ηλεκτρονικών υπογραφών που θα συνάδουν με αυτά τα τεχνικά πρότυπα. Κατά τη γνώμη μα, χρειάζεται υποδομή ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη για όλων των ειδών τη υπηρεσία πιστοποίηση. Μόνο έτσι θα βελτιώσουμε με τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ε, ειδών ηλεκτρονικών υπογραφών. Promotional and educational measures. Χρειάζεται επίσης επικοινωνιακή δράση για την προώθηση τη εννοιά των ηλεκτρονικών υπογραφών. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει για φέτος πρόταση αναθεώρηση οδηγίε για τι ηλεκτρονικέ υπογραφέ, Άρα φαίνεται να τίνει προ την προσέγγιση ευρεία κλίμακο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπροσθέτως και εκ παραλίλου θα θέλαμε να αναλυθούμε τα εξή μέτρα οι φυστάμες ε, Πρωτοβουλίε εναρμόνισης καθώ και τα πιλωτικά προγράμματα που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω το ΠΕΒΛ και το SPOX, πρέπει να συνεχιστούν ε, στην γραμμή τη αναθεωρημένη, του σχεδίου μάλλον αναθεώρηση τη οδηγία. Και μελλοντικά για την ηλεκτρονική αναγνώριση θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω βήματα, διότι η ηλεκτρονική αναγνώριση είναι προπόθεση συχνά ε, για την για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Ε, επίσης, ε, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω οικονομική στήριξη των μέτρων, όπως ε, φορολογικά κίνητρα για τους χρήστες, ώστε να χρησιμοποιούν ευρύτερα τις ηλεκτρονικές υπογραφές, καθώς και κίνητρα για τους παρόχους, ούτως ώστε αυτοί να προσφέρουν τεχνικές και οικονομικές λύσεις και εφαρμογές που θα καλύπτουν το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Αυτές είναι οι συστάσεις μας. Ελπίζω να ήταν πλήρη η παρουσίασή μου σχετικά με τι εξελίξει και τι δράσει που κρίνουμε σκόπιμε στον τομέα των ηλεκτρονικών υπογράφων. Προφανέστατα, αν θέλετε και άλλε πληροφορίε μπορείτε, σας παραπέμπω στην μελέτη μα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σα, κυρίες και κύριοι, και θα δώσω και πάλι το λόγο στη συνάδελφό μου, που θα συνεχίσει με την παρουσίαση του δεύτερου τμήματο τη μελέτη σχετικά με τι ηλεκτρονικέ προμήθειε. Ευχαριστούμε για τον τομέα των ε, ηλεκτρονικών ε, διαγωνισμών είναι σαφές ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ε, τομέας με... για ολόκληρη την οικονομία της Ένωσης για να υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες πιο αποτελεσματικές λειτουργίες οι οποίες δεν γίνονται αυτή τη στιγμή στο βέλτιστο επίπεδο και στον τομέα της διαφάνειας και στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Τα μέτρα αυτά και εδώ πέρα συμφωνούν οι μελέτε θα οδηγήσουν σε πάρα πολύ σημαντική μείωση του κόστους. Όταν μιλάμε για ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών ε, προμηθειών, το... οι δυνατότητες που φαίνεται ότι υπάρχουν είναι πάρα πολύ μεγάλες για εξοικονόμηση κόστους. Αυτό δεν είναι τίποτα το καινούριο. Από το 2004 με το σχέδιο δράσης οι ηλεκτρονικές ε, προμήθειες ε, προβλέπονταν και είχε συντακτική σχετική οδηγία. Πριν ε, περάσουμε στα συγκεκριμένα σημεία, να σας πω τι εννοούμε ηλεκτρονικές προμήθειες. Εννοούμε μια διαδικασία η οποία σε κάποιες ή πιθανώ σε όλες τις φάσεις ε, της ε, προμήθειας βασίζεται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέσω διαδικτύου. Ήδη από τη φάση της προετοιμασίας γνωρίζουμε τις φάσεις. Έχουμε την ηλεκτρονική κοινοποίηση, την αναγγελία του διαγωνισμού, αλλά ακόμα και στη φάση της διεξαγωγής ε, του διαγωνισμού και της αξιολόγησης ε, υπάρχουν ε, ηλεκτρονικές διαδικασίες. Οπότε όταν μιλάμε για αυτό το οποίο απαιτείται ως ελάχιστο για ηλεκτρονικές προμήθειες, μιλάμε για τις τρεις πρώτες φάσεις, ε, δηλαδή ηλεκτρονική προκήρυξη, ηλεκτρονική πρόσβαση και ηλεκτρονική υποβολή, για να θεωρήσουμε ότι έχουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Και εκεί πέρα ακριβώς έχουμε τα περισσότερα προβλήματα όσον αφορά την φάση της υποβολής, γιατί θα πρέπει βεβαίως να είναι πάρα πολύ έντονη η συνεργασία μεταξύ αυτού που προκυρήσει το διαγωνισμό και αυτών που υποβάλλουν ε, προσφορές και η ηλεκτρονική υπογραφή εδώ πέρα παίξει κάποιο ρόλο. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. <coughs> Τι έχει γίνει τώρα στην ε, πράξη όσον αφορά τις προμήθειες στα κράτη-μέλη και πού και αν υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης. Η Πράσινη Βίβλος του 2010 έκανε μια γενική έρευνα βασισμένη σε πάρα πολλές ε, μελέτες. Ε, υπήρχε η μελέτη Siemens Timelex με πάνω από 100 σελίδες και αναφέρονταν εκεί πέρα πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες στα κράτη-μέλη σήμερα. Παρόλα αυτά, παρόλες τις ε, πολλές εργασίες που έχουν γίνει από διάφορα Ινστιτούτα και Ιδρύματα προβληματικό είναι πως ε, πάρα πολλά στοιχεία δεν μπόρεσαν να δοθούν, ειδικά όσον αφορά τις ε, διαγωνισμούς ε, που ήταν κάτω από ένα ορισμένο κατόφλι για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια, αποτε... κάποια αποτελέσματα τα οποία θα είναι αντιπροσωπευτικά. Ποιε είναι λοιπόν οι δυσκολίε σε σχέση με τι χώρε που δεν έχουν προχωρήσει τώρα σε σχέση με αυτά τα οποία φανταζόμασταν το 2004 υπάρχουν όντως ε, κάποιες ε, αμφιβολίες για τη χρήση των ηλεκτρονικών προμηθειών. Όχι, από ό,τι φαίνεται πως υπάρχουν, υπάρχουν μόνο ωφέλη από τις ηλεκτρονικές ε, προμήθειες καθώς είναι κάτι πολύ απλούστερο να γίνει και διασυνοριακά και πιο, να είναι πιο διάφανες οι προμήθειες σε σχέση με την έγγραφη διαδικασία, ειδικά όσον αφορά την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ε, της ε, διαφθοράς μισχόρτα, υπάρχουν πάρα πολλά πλέον εκτήματα. Και βεβαίως υπάρχει η απόλυτη καταγραφή του πώς ε, κινήθηκε το σύστημα. Όσον αφορά λοιπόν την εφαρμογή, νομίζω πως θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο μέλλον σε μια διαδικασία προμηθειών χωρίς χαρτιά και τέλος, ειδικά όσον αφορά την ε, υλοποίηση της ε, σύμβασης ε, νομίζω πως μπορούμε να οδηγηθούμε σε καλύτερες τιμές και σε πιο γρήγορη πληρωμή των αναδόχων του έργου. Τώρα, ποια είναι τα πιθανά μειονεκτήματα. Αυτά διαπιστώνονται μόνο εκεί όπου δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών προμηθειών. Μία πτυχή που διαψώνουμε ήδη εκεί όπου έχουν εφαρμοστεί ηλεκτρονικές προμήθειες είναι πως ε, λόγω των απαραίτητων ικανοτήτων που χρειάζονται κυρίως κεντρικές υπηρεσίες ε, σε κράτη-μέλη που το εφαρμόζουν όπως παραδείγματο χάρη στην ε, Αυστρία Ε, βλέπουμε πως μπορούμε να ε, μπορούν, πρέπει να λειτουργήσουν ε, εντός ενός πλαισίου αλλά βλέπετε πως το πλαίσιο αυτό το οποίο έχουν ίσως να εμποδίζουν ως ένα βαθμό τον ανταγωνισμό. Και βεβαίως η διαδικασία Πηγαίνετε στην προηγούμενη διαφάνεια αν θέλετε. Κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε στην πράξη ως ε, μειονέκτημα είναι πως η διαδικασία της αξιολόγησης ειδικά σε πολύπλοκα έργα δεν είναι πάντα κάτι το υπολογίσιμο με μαθηματικούς τύπους, ειδικά όταν υπησέρχονται ποιοτικά κριτήρια και άρα βλέπουμε πως ε, απομακρύνονται από αυτά ειδικά τα κριτήρια οι χρήστες και επικεντρώνονται ξανά μόνο στην τιμή και άλλα μετρήσιμα κριτήρια, κάτι το οποίο δεν είναι οπωσδήποτε ε, πάντα θετικό. Και επίσης έχουν δυσκολία οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να περάσουν στις ηλεκτρονικές προμήθειες γιατί χρειάζεται βέβαια μια αρχική επένδυση για να εξοικειωθούν και με το σύστημα. Λοιπόν, επόμενη διαφάνεια. σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη υπάρχει νομική βάση, βάση για την ε, χρήση των ηλεκτρονικών ε, προμηθείων. Δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη διαμορφώσει όλες τις φάσεις των ηλεκτρονικών ε, προμηθειών. Υπάρχουν όλες οι φάσεις από μια πρώτη γνωριμία μέχρι ολοκλήρωση του συστήματος. Βλέπετε πως γίνεται κάποια διάκριση στο πλαίσιο των νομικών βάσεων εδώ πέρα που υπάρχει. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά εάν δείτε το εύρος της πρακτικής ε, όσον αφορά πέρα από το νομικό πλαίσιο την πραγματική εφαρμογή. Υπάρχουν κάποια κράτη πρωτοπόροι όπως η Πορτογαλία που έχει προχωρήσει πάρα πολύ στις ηλεκτρονικές ε, προμήθειες καθώς για συγκεκριμένες προμήθειες είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διεξαγωγή και οι μελέτες δείχνουν πως υπάρχουν ήδη αποτελέσματα. Στην ε, Πορτογαλία 75% όλων των προμηθειών πλέον είναι ηλεκτρονικές και αυτό έχει οδηγήσει σε μια εξοικονόμηση 10 έως 20% και μια εξοικονόμηση του διοικητικού κόστους κατά 60%. Και άρα στην εφαρμογή στα κράτη-μέλη υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα, αλλά είναι τεράστιο το φάσμα, βλέπετε, μεταξύ των κρατών μελών. Επόμενη διαφάνεια. Και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πάρα πολλές ε, υποστηρικτικές ε, πρωτοβουλίες ε, σε διάφορα στοιχεία των ηλεκτρονικών προμηθειών. Τα ανέφερε ήδη η κυρία Χόφμαν το ΠΕΠΟΛ παραδείγματο χάρη έχει μια συνολική προσέγγιση, έχει κάποια συστατικά που μπορούν να απτυχθούν αμέσως ε, θα λέγαμε και μετά με βάση αυτά τα έτοιμα κομμάτια μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια πλήρη ηλεκτρονική ε, προμήθεια που θα λύνει πολλά προβλήματα στις διασυνοριακές ειδικά προμήθειες. Το e-cert της παραδείγματος χάρη είναι ένα μέσο πληροφόρησης ε, και για τις παραδοσιακές θα έλεγα προμήθειες καθώς διευκολύνει την πληροφόρηση και άλλων κρατών μελών. Οπότε συμβαίνουν πάρα πολλά αυτή την στιγμή και οπωσδήποτε δεν έχουμε επιτύχει αυτό το οποίο ελπίζαμε το 2004. Στην επόμενη διαφάνεια περνάμε στα εμπόδια τα οποία συναντήσαμε και στα οποία οφείλεται η κατάσταση. Τα βασικά εμπόδια τα οποία συναντήσαμε είναι το ότι δεν υπάρχουν ενιαίες ε, αποδεκτές πορδιαγραφές, ειδικά στο τεχνικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλές μεμονωμένες λύσεις. Το πρόβλημα αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ομοσπονδιακά κράτη-μέλη και ειδικά στη Γερμανία διαπιστώνουμε πως υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις ε, και κάποιες ακολουθούνται μόνο σε ένα δήμο παραδείγματο χάρη και μόνο τώρα γίνεται η προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο μέσω μιας κεντρικής υπηρεσίας να υπάρχει ένας συντονισμός να προσφερθούν έτσι εργαλεία για λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αφορά και τις παραδοσιακές ε, προμήθειες αλλά μας δίνει την δυνατότητα και μας ε, δίνει βεβαίως ε, μας δείχνει την ανάγκη να καταλήξουμε σε κάποια αισθήματα είναι και το γλωσσικό ε, φράγμα. Όλα αυτά βεβαίως τα εμπόδια έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα στις διάφορες φάσεις της προμήθειας. Όσον αφορά παραδείγματος χάρη την πρόσβαση στους φακέλους διαπιστώνουμε πως όσον αφορά την τεχνική πρόσβαση υπάρχουν κάποια εμπόδια, αλλά εξαρτάται από το πόσο πολύπλοκη είναι η τεχνική λύση η οποία έχει ακολουθηθεί. Υπάρχουν παραδείγματο χάρη σχετικά απλέ λύσει για πρόσβαση που ζητάνε μόνο μια καταγραφή και ένα συνθηματικό, αλλά ειδικά όσον αφορά τις ε, διασυνοριακές ε, προμήθειες ε, υπάρχουν προβλήματα ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα όμως τα προβλήματα υπάρχουν στην φάση της υποβολής των προσφορών. Εδώ πέρα υπάρχει πάλι το ζήτημα της γλώσσας και εδώ πέρα υπάρχει πάλι το ζήτημα του ότι οι διάφορες ε, λύσεις που έχουν υιοθετηθεί διαφέρουν πάρα πολύ. Αυτό αφορά το θέμα της ταυτοποίησης του χρήστη. Ξέρετε πως αυτά τα ακούσαμε και στο θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής. Να εξηγήσω περί την πρόκειται. Το θέμα είναι δηλαδή ποιος είναι αυτός που υποβάλλει την προσφορά και πώς μπορώ να διασφαλίσω πως ε, πράγματι η δήλωση, η υποβολή προσφοράς που βλέπω εδώ πέρα είναι δική του. Οι δε σχετικές οδηγίες ε, έχουν ε, ορίσει πάρα, πολλούς λίγους κανόνες, πάρα πολύ λίγους κανόνες σε αυτόν τον ε, τομέα. Δεν υπάρχει κάποια απέτηση, παραδείγματο χάρη, για ένα σύστημα υπογραφών. Οπότε οι οδηγίες περί προμηθειών λένε μόνο πως θα πρέπει να φτάσει μυστική η προσφορά. Ζήτημα ταυτοποίηση και υπογραφών δεν αναφέρεται. Οπότε στο θέμα της υποβολής των προσφορών και το πώς θα πρέπει να συμβεί υπάρχει πάρα πολύ, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν μοντέλα όπως στην Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία που έχουν ε, ένα σχετικά απλό σύστημα με ένα όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό για την ε, ταυτοποίηση αυτού που υποβάλλει τις ε, προσφορές. Επίσης ε, πάρα πολλά άλλα κράτη-μέλη όπως η Γερμανία, η Αυστρία εργάζονται με λύσεις υπογραφής και εδώ πέρα έχουμε το πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε πριν πως ε, υπάρχει το ζήτημα της αποδοχής ειδικά όσον αφορά κάποιους από άλλα κράτη-μέλη και πρόβλημα συμβατότητας. Πέρασε παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια. Όσον αφορά τον τομέα της ε, εξέτασης ε, της ταυτοποίησης όπως σας είπα δηλαδή το πώς ε, θα μπορέσουμε και να δούμε τι αξία και τι περιεχόμενο έχουν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από κάποιο άλλο κράτος μέλος. Γιατί βλέπετε άλλα κράτη-μέλη απαιτούν μόνο το πρωτότυπο με υπογραφή κτλ. Και εδώ πέρα μπορούν να υπάρξουν πολλές βελτιώσεις. Τέλος, όσον αφορά την ε, τιμολόγηση, υπάρχουν ε, λόγω ακριβώς των νομικών διαφορών στα κράτη-μέλη. Υπάρχει και πρόβλημα βεβαίως ε, αποδοχής γιατί υπάρχουν ε, ανησυχίες για ε, νομικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Και όπως σας είπα διαφέρουν οι διαδικασίες στα κράτη-μέλη. Τώρα, αν περάσουμε σε μη πρωτότυπες λύσεις, αλλά όπως σας είπα σε κάποια υποδείγματα ηλεκτρονικών προμηθειών, έχουμε το θέμα του, ε, των ε, συμφωνιών πλαισίων ε, και συχνά συνδέεται βεβαίως η ηλεκτρονική προμήθεια με μια κεντρική υπηρεσία. Βεβαίως ε, το ζήτημα είναι πως μετά έχουμε τρία-τέσσερα χρόνια ένα κλειστό σύστημα το οποίο δεν επιτρέπει ένα άνοιγμα στην αγορά για να επιτρέψει τη συμμετοχή και άλλων επιχειρήσεων. Οπότε αυτό αντιμετωπίζεται με ένα δυναμικό σύστημα προμηθειών ε, το οποίο μας επιτρέπει να περάσουμε στον ηλεκτρονικό κόσμο, αλλά πρέπει να πούμε πως η αποδοχή του δυναμικού συστήματος προμηθειών μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί η χρήση και στο τεχνικό επίπεδο ενός τέτοιου συστήματος ε, σημαίνει πάρα πολύ μεγάλες αρχικές ε, επενδύσεις και έξοδα. Μας ρώτησαν ειδικά το τι θα πρέπει να γίνει τώρα με τα πολύ ε, κρίσιμα σημεία της υποβολής των προσφορών και της ταυτοποίησης ε, ε, αυτών οι οποίοι υποβάλλουν τις προσφορές. Εδώ πέρα βλέπουμε πως πρέπει να υπάρξει να γίνει πραγματικά κάτι, ειδικά όσον αφορά την διασυνοριακή λειτουργία. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι πως στην χρήση ηλεκτρονικών ε, υπογραφών αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια νομικά ασφαλής ε, λύση γιατί δεν είναι υποχρεωτικά, υποχρεωτικό ακόμα να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής ε, υπογραφής μπορούν να ακολουθηθούν παραδείγματος χάρη τα μοντέλα της Ιρλανδίας όπως σα είπα με ένα όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό αλλά θα έπρεπε νομίζω ως ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας να υπάρξει ένα token το οποίο μπορεί κανείς να κατεβάσει στο σύστημά του ακριβώς για να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στο σύστημα και αυτό βεβαίως σημαίνει λιγότερες δυσκολίες όσον αφορά διαλειτουργικότητα, γλωσσικά ζητήματα κτλ. Και νομίζω μπορεί να οδηγήσει στα κάρτα εκείνα στα οποία χρησιμοποιείται σε πολύ μεγαλύτερη αποδοχή. Επόμενη διαφάνεια. Τα επόμενα βήματα, τα οποία κατά την άποψή μας θα είναι σωστά, είναι να συνεχίσουμε τα καλά έργα τα οποία υπάρχουν, αλλά πολλά από αυτά χρηματοδοτούνται και είναι παράλληλα. Ειδικά το ΠΕΠΛ e έχει νομίζω πάρα πολύ καλές προοπτικές και ένα συντονισμός αυτών των έργων θα μπορούσε σύντομα να φέρει τα πράγματα σε ένα επόμενο επίπεδο για να οδηγηθούμε σε πολύ πιο ε, διαδεδομένη χρήση στην πράξη. Δεν θα πρέπει να προσθέσουμε νέες προδιαγραφές σε αυτές οι οποίες ήδη υπάρχουν θα πρέπει νομίζω να κινηθούμε στο πλαίσιο των υπαρχών αισθημάτων να μην υπάρξει κι άλλος ε, κατακαιρματισμός. Τώρα, αυτά τα οποία ακούστηκαν περί υποχρεωτικών ηλεκτρονικών προμηθειών δεν θα πρέπει νομίζω να συνδεθούν με μία προθεσμία και μία λύση η οποία θα επιβληθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ε, δοθεί μια κάποια όθηση οπωσδήποτε, αλλά πάντα στο πλαίσιο μιας εναρμόνισης ε, για να μπορέσουμε να πάρουμε μαζί μας ε, και τους ε, αναδόχους, γιατί συχνά υπάρχουν ειδικέ υπηρεσίες για τις προμήθειες που έχουν αρκετά εκτεταμένη τέχνογνωσία, αλλά ασχολούνται και με πάρα πολλά ε, άλλα ζητήματα, όχι μόνο με τις προμήθειες. Οπότε οι χρήστες θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδεχτούν τις νέες λύσεις για να οδηγηθούμε σε κάποια αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων αυτών σε αυτά τα υποστηρικτικά νομίζω μέτρα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία καλό θα ήταν να προσθεθεί να δούμε και κάποιες διευκρινήσεις στην οδηγία περί προμηθειών πρώτα απ' όλα υπάρχουν ήδη κάποιες ε, αμφιβολίες για το εάν θα μπορούσε να αποτελήσει διακριτική μεταχείριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η ηλεκτρονική προμήθεια Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται περί θεμητής λύσης που δεν έχει. Μετά να δούμε το τι θα γίνει και θα πρέπει να μπορέσουμε να εργαστούμε με δηλώσεις από πλευράς των ιδίων των αναδόχων και να μην αναζητούν πάντα πιστοποιητικά από τις αρχές. Βεβαίως θα πρέπει πάντα να έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αργότερα στην διαδικασία της βεβαιώσεις αυτές, αλλά κατά τη διάρκεια της ε, προμήθειας ε, θα μπορούσαμε να περιοριστούμε σε μία δήλωση του πιθανού αναδόχου. Και βεβαίως υπάρχει δυνατότητα, όπως σας είπα, για το δυναμικό σύστημα προμηθειών, το οποίο θα διευκόλυνε τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και τώρα είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Euh, να δώσω το λόγο. Άντε, αν θέλει να πει κάτι για τις δημόσιες προμήθειες, καλό θα είναι να ακούσουμε την άποψη της ε, καθώς είναι συγκήτρια. Σύντομα, γιατί για να πω την αλήθεια δεν μας είπατε και τίποτα το καινούριο. Εγώ τα ήξερα αυτά. Οπότε για εμένα ενδιαφέρον είναι να ενσωματωθούν οι ηλεκτρονικές προμήθειες στην αναθεώρηση της οδηγίας περί προμηθειών. Για εμένα επίσης ε, δυστυχώς δεν αναφέρθηκε στη μελέτη το ότι η Κομισιόν πρέπει να επιδείξει περισσότερη πολιτική ηγεσία και να αναλάβει περισσότερη πολιτική ευθύνη και να γίνουν συμβατές οι διάφορες πλατφόρμες ε, που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δυσκολεύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και κατά τα λοιπά τα υπόλοιπα τα στηρίζω για ευκολότερη πρόσβαση. Πράγματι δεν καταλαβαίνω γιατί ε, μια ηλεκτρονική προμήθεια είναι υψηλότερο εμπόδιο από μια προμήθεια με χαρτιά. Αλλά βεβαίως πρέπει να πούμε, το είπατε στην ηλεκτρονική υπογραφή και με τις χρονικές σφραγίδες, υπάρχουν προδιαγραφές που δεν είναι εναρμονισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εναρμονίσει αυτές τις προδιαγραφές και να προτείνει ανοιχτά φόρματ ε, τα οποία θα είναι και τεχνολογικά ουδέτερα. Νομίζω πως είναι σημαντικό αυτό. Αλλά θα ήθελα να τα συμπεριλάβω αυτά στην ε, έκθεσή μου, αλλά υπάρχει βεβαίως το ζήτημα της ε, συντομίας του περιορισμού μεγέθους της έκθεσης θα μπορούσαμε να καταθέσουμε τις ηλεκτρονικές προμήθειες ως τροπολογία να κάνουμε κάποιο κόλπο εκεί πέρα. Ούτως ή άλλως θα τα στείλω εκ των προτέρων και στα αγγλικά για να μπορέσετε να καταθέσετε τροπολογίες. Ευχαριστώ. Θα έλεγα απλώ ότι συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σα. Πρόκειται για μια αναγκαιότητα. Πρέπει να ε, επικαιροποιήσουμε και εμεί τη θέση μα ανάλογα με τον 21ο αιώνα. Πάρμπαρα. Ναι. Τα καλά παραδείγματα τα οποία αναφέρατε της Ιρλανδίας, της Αυστρίας, της Εσθονίας, Πορτογαλίας, οπωσδήποτε ε, να τα υιοθετήσουμε. Ελπίζω η Κομισιόν να ήταν παρούσα και να σημείωσε τις προτάσεις αυτές για τις τεχνικές βελτιώσεις για τις οδηγίες, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει... Βεβαίω είναι πολιτικό το ερώτημα, παρόλα αυτά θα το θέσω όσον αφορά την, ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αυτά τα οποία έχετε πει ως ε, χρήση συγκρούνται με τις πολιτικές μας ιδέες, δηλαδή ποια κριτήρια θα πρέπει να προωθήσουμε, να στηρίξουμε για να εμπλακούν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ό,τι μέχρι τώρα. Οπότε το ερώτημά μου είναι πώς θα μπορέσετε με τις τεχνικές προτάσεις σας να μας δώσετε μια ιδέα για το πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πολιτικό ζήτημα και να το θέσουμε και στον Επιτρόπο Μπαρνιέ. Πώς θα τα συμβάσουμε όλα αυτά με τα τεχνολογικά δεδομένα. Από ό,τι καταλαβαίνω, νομίζω πως αυτό είναι δυνατόν Όπω σας είπα, το θέμα δεν είναι τόσο τα πλεονεκτήματα, είναι τα μειονεκτήματα, είναι η μη σωστή εφαρμογή, γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολύ μεγάλες, ε, πάρα πολλά, να έχουμε πάρα πολλά μεγάλα ωφέλη και στις πρώτες φάσεις, αλλά και στη διαδικασία της αξιολόγησης, ε, να ξαναπάμε λίγο πιο, πολύ, πιο κοντά στο φυσιολογικό κόσμο για τα μαλακά αυτά σας είπα τα μη ε, μετρήσιμα τόσο κριτήρια τα οποία μπορούν να ληφθούν ε, ως ε, όχι ε, κάτι το επιπρόσθετο αλλά ως κάτι το επίσημο να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία μπορεί να απαντηθούν ξέρω εγώ το εκπληρώνει ναι όχι οπότε νομίζω μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο βεβαίως μετά δεν θα μιλάμε για ηλεκτρονική προμήθεια από το α ως το ω θα υπάρχει στη διαδικασία της αξιολόγησης μια διακοπή ε, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε πράγματι αν εκπληρώνονται κάποια από αυτά τα κριτήρια. Αλλά αυτό δεν είναι εμπόδιο στην ε, χρήση των ηλεκτρονικών προμηθειών. Απλά δεν είμαστε από το α στο ω χωρίς χαρτιά εάν θέλετε, σε ηλεκτρονική μορφή. Απλά επισέρχεται κάπου το, επισέρχονται κάπου αυτά τα ποιοτικά τα κριτήρια. Τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό το συμπεριλάβαμε στην ε, μελέτη. Νομίζω στη Δανία, παραδείγματο χάρη, ε, υπάρχει ήδη πάρα πολύ ηλεκτρονική τιμολόγηση. Υπάρχει μία κεντρική υπηρεσία η οποία ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει και τους εξηγεί πως από εδώ και μπρος τα τιμολόγια αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά και στηρίζει πραγματικά την εφαρμογή του των νέων αυτών εντό εισαγωγικών ε, μεθόδων, ειδικά όσον αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι στη διάθεσή του. Και εδώ πέρα ακριβώς είναι το ζήτημα των υποστηρικτικών μέτρων, γιατί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω συνδέσμων επιμελητηρίων ε, μπορούν να έχουν έναν ε, συνομιλητή για να τους δείξει πώς έχουν τα πράγματα και νομίζω πως ε, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ απλώστερα εάν μειωθούν ορισμένα εμπόδια όπως παραδείγματο χάρη αυτό της υπογραφής αυτομάτως θα γίνει πολύ ευκολότερη κατάσταση για τις ε, μικρόμεσαίες επιχειρήσεις. Ε, νομίζω ότι για να διεξαχθεί εύρυθμα η συζήτηση ε, καλό είναι να ακούσουμε τους βουλευτές και θα σας ξαναδώσουμε το λόγο στη συνέχεια γιατί μην ξεχνάτε ότι θα ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν ακούσουμε την κυρία Στίτλερ, θα ήθελα να καλωσορίσω από πλευρά του Hans Πίτερ Mayer μια ομάδα επισκεπτών καλωσορίσατε στη συνεδρίασή μας και ελπίζω ότι θα αποκομίσετε μια θετική εντύπωση για τις εργασίες της Επιτροπής Οστερικής Αγοράς που είναι και μια από τις σημαντικότερες του Κοινοβούλιο. Κάτριν. Thank you. Um, ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Μόλις μας είπατε ότι για τις προμήθειες ε, υπάρχει θέμα επαγγελματισμού, δηλαδή θέμα εφαρμογής των κανόνων και υπάρχουν νέες προκλήσεις για τις ηλεκτρονικές ε, προμήθειες. Θα μπορούσατε ίσως να εμβαθύνετε Επίσης, ε, στην παρουσίαση είπατε κάτι ενδιαφέρον. Μιλήσατε για την εμπιστοσύνη. Μέχρι να εμπιστευτούν το σύστημα οι χρήστες, δεν πρόκειται ε, να ακολουθήσουν το καρότο. Δηλαδή, όταν δίνουμε κίνητρα για να αρχίσει κάποιος να χρησιμοποιεί το σύστημα, ίσως δεν επαρκεί. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας ίσως. Μιλήσατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, παραδείγματος χάρη. Ε, και σε σχέση με πώς επηρεάζει η δράση τους ε, το όλο θέμα. Φυσικά είναι σημαντικό, φυσικά είναι καταλητικός ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία και μπορούν να μας ε, βοηθήσουν οι επιχειρήσεις να καταλάβουν τα περί απροθυμίας ως προς τη χρήση του νέου συστήματος. Μα είπατε επίσης ότι υπάρχουν προκλήσεις διότι τα κράτη-μέλη λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Εμείς στη Σκοτία, παραδείγματος χάρη, από την εκχώρηση της εξουσίας σε περιφερειακό επίπεδο αλλάξαμε άρδιν το σύστημα για τις ε, προμήθειες και άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνη και συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, μια διασυνοριακή συνεργασία για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τι βέλτιστε πρακτικέ και να αποκομίσουμε τα μάλλα από το νέο σύστημα. Στην παρουσίαση μα είπατε ότι το 19% είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί στι ηλεκτρονικέ προμήθειε. Και άρα προετοιμά, ε, αναμένοντας ε, την πράσινη βίβλο και την επόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να μελετήσουμε όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσετε τις βέλτιστες πρακτικές που αναφέρατε κι εσείς ε, στην παρουσίασή σας και επίσης πώς βλέπετε τις μελλοντικέ προοπτικές των ηλεκτρονικών προμηθειών. Ευχαριστούμε Κατρίν Πρόεδρος. Η Χάιντι έχει ξαναστήσει το λόγο. Συγγνώμη να αναφερθώ στο ερώτημα της κυρίας Βάιλερ. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω πως πρέπει να είναι υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές προμήθειες και δεν θεωρώ πως μπορούν να αντικαταστήσουν τα πάντα. Να το ξεκαθαρίσω αυτό γιατί υπάρχουν και άλλες μέθοδοι όπως η διαδικασία της διαπραγμάτευσης που είναι εξίσου αποτελεσματική αν μιλάμε για καινοτόμες μεθόδους οι ηλεκτρονικές προμήθειες έχουν πλεονεκτήματα για τυποποιημένα προϊόντα, για απλές διαδικασίες. Εκεί πέρα έχει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα και οπωσδήποτε βλέπετε πως έχουμε μόνο ένα 5% τις των προμηθειών που γίνονται ηλεκτρονικές ενώ η Κομισιόν ήθελε να φτάσουμε ε, το 50. Δεν θα αντικαταστήσει λοιπόν όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Ευχαριστώ. Καθώς μας μένουν μόνο πέντε λεπτά, θα δώσω μέσο στο λόγο στην κυρία Καναλοπούλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκαμε Σάνκο. Uh, Γεια σας, ε, δεν ζήτησα το λόγο. Ε, εκπροσωπώ τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ, αλλά δεν είμαστε καθήλυνα αρμόδια γενική διεύθυνση. Δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε προς το παρόν. Μάλιστα, εφόσον δεν υπάρχουν σχόλια από την πλευρά της Κομισιόν. Α, υπάρχει κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί εξ όνομα της Κομισιόν, μάλιστα. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Λέγομαι Γκαλέρ ε, και είμαι policy officer αρμόδιος ε, για την ε, Οδηγία για τις ηλεκτρονικές επιγραφές. Ε, ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που μας ε, κάλεσε εδώ να λάβω σημειώσεις. Αυτό έκανα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ε, διάβασα και την έκθεση και θεωρώ ότι πράγματι παρουσιάζει με σύνθετο τρόπο τη δουλειά που κάνουμε εδώ και κάποια χρόνια. Καλό λοιπόν όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαβάσουν την έκθεση. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διευκρίνηση ότι ορισμένα νέα στοιχεία ουσιαστικά συνδυάζονται με ε, μια νέα μελέτη που αφορά την ε, ηλεκτρονική υπογραφή και την ε, ταυτοποίηση της αυθεντικότητας της υπογραφής. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτά τα νέα στοιχεία. Μάλιστα, ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι, θα ολοκληρώσουμε λοιπόν εδώ τη συζήτηση και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο σε δύο λεπτά. Λοιπόν, παρακαλώ όσοι είναι να εγκαταλείψουν την αίθουσα να το κάνουν με ησυχία και γρήγορα. Σας παρακαλώ και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει μια παρουσίαση της ε, λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Καταναλωτικών Κέντρων ε, μετά από πέντε έτη. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό τον απολογισμό θα δώσω το λόγο στον ε, επικεφαλή τη Διευθύνση ε, τη ΓΔ τον κύριο Στάμα Μολνάρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να καλωσορίσω και τους αξιότιμους κύριους βουλευτές, τους επικεφαλής και όλους τους υπολοιπούς που αποφάσισαν να, να παρευρεθούν σε αυτή την παρουσίαση. Όπως αναφέρατε, το δίκτυο ECC πέρσι ολοκληρώσε το πέμπτο έτος ε, ύπαρξής του, η Κομισιόν ε, αποφάσισε να προβεί σε μια διαδικασία αξιολόγηση. Βλέπετε εδώ στην εικόνα τα μέλη, τους διευθυντές ε, του ECCNet, του δικτύου αυτού των κέντρων καταναλωτών και μπορεί να δείτε και ανθρώπους που γνωρίζετε σε αυτή τη φωτογραφία και η Επιτροπή αυτή, καθώς γνωρίζει πολλά για το δίκτυο, θα κάνω μια σύντομη σύνοψη σε τι συνιστά το δίκτυο και τι συμβαίνει. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο. Έχουμε γραφεία σε κάθε κράτος μέλος και στην Ορδηγία και στην Ισλανδία. Και περατώντας αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του δικτύου είναι να ενημερώσει και να υποστηρίξει τους καταναλωτές, ε, οπότε ε, συμμετέχουν σε κάποια διασυνοριακή δραστηριότητα. Παραδείγματο χάρη, ε, όποτε επισκέπτονται κάποια άλλη χώρα και αγοράζουν κάτι, μπορούν να στραφούν στα ICC. Θέλω να ανακοινώσω ότι το 2010 τα κέντρα ε, καταγράψαν πάνω από 70.000 επαφές με τους καταναλωτές ε, και ε, αυτό συνιστά πολύ μεγάλη γνώση και από τη στιγμή που ξεκίνησε το δίκτυο το 2005 καταγράψε 340.000 επαφές. Προϋπολογισμός που χρησιμοποιήσαμε συνολικά τα κρατη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 8,6 εκατομμύρια το χρόνο. Και αν δείτε τη διαφάνεια, βλέπετε τον ε, αριθμό των περιπτώσεων, έχουμε αύξηση χρόνο με το χρόνο αριθμό των υποθέσεων. Τώρα, σε αυτή τη διαφάνεια στην οθόνη βλέπετε τους τομείς ε, όπου παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα, δηλαδή για τις οποίε υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες. Ε, κυρίως έχουμε καταγγελίες για τις μεταφορές, ε, δεύτερο το τομέα ανεψυχής και κατόπιν εστιατόρια και ξενοδοχεία. Αυτή είναι οι τρεις κύριοι τομείς ε, όπου υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Αν δείτε την μέθοδο πώλησης, ε, πρώτο βρίσκεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και ε, το δεύτερο είναι μόνο το 1 τρίτο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι διασυνορικές δραστηριότητες που γνωστοποιούνται στο ΙΣΣΥ αφορούν κυρίως δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου. Και τώρα φτάνουμε στη διαφάνεια που αφορά την εξωτερική αξιολόγηση. Η Κομισιόν αποφάσισε να ξεκινήσει μία εξωτερική αξιολόγηση για δύο λόγους. Καταρχήν, για να αξιολογήσει τη λειτουργία του δικτύου μέχρι σήμερα και να έχουμε δεύτερον μία εξωτερική εικόνα από κάποιον εξάρτητο φορέα και αναμέναμε να προκύψουν και κάποιες συστάσεις για το μέλλον. Θα ήθελα να υπογραμμίσω στο στάδιο αυτό ότι η μελέτη και τα πορίσματα δεν ε, είναι επίσημα πορίσματα της Κομισιόν. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν και το τρίζεται εδώ η άποψη του συγκεκριμένου φορέα. Στην ε, επόμενη διαφάνεια συνοψίζουμε τη διαδικασία. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Ξέρω ότι είμαι το τελευταίο εμπόδιο μεταξύ μόνο και του γευματό σα. Έτσι λοιπόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε και αν έχετε φυσικά ερωτήσει θα επανέλθουμε. Έτσι λοιπόν, στην αρχή αυτού του έτου. λάβαμε την τελική έκθεση. που προσπαθούσε να απαντήσει στα εξή ερωτήματα. Εδώ το ομοδοποιούμε. Αυτή η διαφάνεια είναι μάλλον η σημαντικότερη σε ό,τι φορά τα ερωτήματα. Έτσι λοιπόν, σχετικότερα και αντίκτυπο ε, του δικτύου, ε, απαντά στι ανάγκε των καταναλωτών, κάποιοι στόχοι ή δραστηριότητε θα πρέπει να προσθεθούν στη λειτουργία του δικτύου, συνεισφέρει το δίκτυο στην επίτευξη των στόχων ε, της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής για τον καταναλωτή και ποιος είναι ο αντίκτυπος σε εθνικό επίπεδο. Προσπαθήσαμε να τα όλα αυτά και να αναφερθούμε στα πλέον σημαντικά ζητήματα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι ορισμένες ρωτήσεις αφορούσαν την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή, την αποδοτικότητα του κόστους, Υπάρχουν ε, κάποιες συστάσεις για βελτίωση επίσης. Ας περάσουμε λοιπόν στη διαφάνεια υπάρχουν 6. Εδώ έχουμε τα κυρία πορίσματα. Καταρχήν, συμπέρανε μελέτη ότι το δίκτυο SSE έχει μια θετική αναλογία κόστος ωφέλους για κάθε ευρώ που επενδύεται στην δραστηριότητα του δικτύου 1,77 ευρώ ε, αξίας 1,77 ευρώ καταγγελίες επιλύονται. Έτσι λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη απόδοση από τις επενδύσεις μας. Υπάρχει και άλλη μια αναλογία για την οποία είμαστε ε, πολύ περήφανοι. Αφορά το μέγεθος ε, των διασυνοριακών ζημιών που, υφίσταται που υφίστανται οι καταναλωτέ εκτιμούμε ότι είναι μεταξύ 500 εκατομμυρίων έως 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίω και το δίκτυο SSC καλύπτει τα 14 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω κάτω μιλάμε μόνο για το 2,3% των αναγκών. Δηλαδή με άλλα λόγια μπορώ να πω ότι ε, περίπου ε, χρειαζόμαστε 30% παραπάνω δραστηριότητα του ΙΣΣΥΜ. Έτσι λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα εδώ και χώρος για βελτίωση. Ο όγκος αυξήθηκε κατά 20% σε 5 χρόνια και αν προσθέσω και το 2010 που δυστυχώς δεν καλύφθηκε γιατί συντάχθηκε η έκθεση κατά το έτος 2010 αυτή η βελτίωση φτάνει το 40% και πιστεύουμε ότι το δίκτυο ECC βοηθά όχι μόνο τους καταναλωτές αλλά και τους εμπερβόμενους, τις επιχειρήσεις γιατί παρέχουμε ίσους κανόνες για όλους, τίθεται κάποια πρότυπα και διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να χαίρουν των δύο δικαιωμάτων σε όλες τις εταιρείε. Υπήρξε και ένα exit poll. Οι χρήστες του δικτύου ΣΥΣΥ ρωτήθηκαν για τη χρησιμότητα του δικτύου και το 87% όσων απάντησαν θεώρησαν ότι η υπηρεσία ήταν χρήσιμη. Αδυναμίες. Δυστυχώς, ε, η γνώση μας για το δίκτυο ECC είναι σχετικά χαμηλή. Μόνο το 15% των πολιτών και 20% των ε, διασυνοριακών αγοραστών έχουν ακούσει το ECC. Φυσικά υπάρχουν κάποιες συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Επίσης, ε, τα κέντρα μας είπαν ότι υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητες ως προς τη χρηματοδότηση ε, το σύστημα χρηματοδότησης είναι ετήσιο και δεν τους επιτρέπει να καταρτήσουν πιο μακροπρόθεσμα σχέδια. Και τέλος υπάρχει ε, το θέμα της ε, προσφυγής. Η, πρόσβαση στις προσφυγές είναι πολύ περιορισμένη γιατί τα ECC δεν μπορούν να, να αναγκάσουν τις εταιρείε να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης και πολύ συχνά οι προσπαθίες τους αποτυγχάνουν. Αν δείτε την επόμενη διαφάνεια, βλέπετε ότι περίπου το 39% των περιπτώσεων δεν επιλύονται γιατί δεν βρέθηκε καμία λύση. Αυτό είναι ο δεύτερος μεγαλύτερο, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό αριστερά και βλέπετε και τι γίνεται με αυτές τις ε, περιπτώσεις, για ποιο λόγο δεν βρέθηκε λόγο. Στο 75% λέγεται ότι οι επιχειρήσεις δεν συνεργάστηκαν, δεν ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για να επιλύσουν το πρόβλημα με τον καταναλωτή. Στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε τα αποτελέσματα της ε, δημοσκόπησης ε, στους καταναλωτές. Βλέπετε εδώ ότι περισσότεροι καταναλωτές που χρησιμοποίησαν το δίκτυο ίσως ήταν πολύ ικανοποιημένοι. Ορισμένοι ήταν ικανοποιημένοι και έχουμε και ένα 11% που ήταν δυσαρεστημένο. Έτσι λοιπόν σκοπεύουμε να συλλέξουμε τέτοιες χρησιμές πληροφορίες και στο μέλλον. Συστάσεις. Και πάλι έχουμε ομάδες συστάσεων, θα τα δούμε εντάχει και βλέπετε κάποιες λεπτομέρειες στη διαφάνεια. Αν έχετε ερωτήσεις, στη συνέχεια θα απαντήσω. Ευχαριστώ. Καταρχήν, η μελέτη αναφέρεται στην πρόθεση ε, και στην ε, ε, προβολή ε, στόχος είναι να συντονιστούν κάποιες, ε, να οργανωθούν κάποιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης αν είναι δυνατό και με άλλους ε, και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εδώ να αναφερόμαστε στι υπουργεία, σε κυβερνήσεις, οργανώσεις καταναλωτών ή όποιον ενδιαφέρεται για να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοδοτική βεβαιότητα, η σύσταση ε, μας προτείνει να χρησιμοποιήσουμε μία τετραετή συμφωνία σύμπραξης ε, με την ε, φιλοξενούσα οργάνωση για να αυξήσουμε τη σταθερότητα και τη συνέχεια επίση ε, προτείνω να χρησιμοποιήσουμε κάποια benchmarks επιδόσεων και επίση κάποια κίνητρα που θα βασίζονται στι επιδόσει. Όμω η Κομισιόν το θεωρεί ότι είναι κάπω δύσκολο γιατί δεν είναι απόλυτα συμβατό με το χρηματοδοτικό κανονισμό. Επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένε συστάσεις για την εσωτερική διαχείριση του δικτύου, απαιτούνται ορισμένα πρότυπα, χρειάζεται κάποια δουλειά για να τεθούν προτεραιότητε, για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση απέναντι στι διάφορες περιπτώσεις και πολύ σημαντικό οι συστάσεις τονίζουν ότι ο ρόλος των θα πρέπει να διευκρινιστεί ως ε, προς τα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ε, των φορέων ε, επιβολής του νόμου και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν εδώ και σε άλλες επιτροπές μπορεί να ακούσετε πολύ, πολύ συχνά το Solvit, το FinMAT. Έτσι λοιπόν πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν τι είναι, τι και ποιος κάνει τι. Αυτό λέμε εδώ, ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στον λόγο τομέα. Σε ό,τι αφορά τη χάραξη πολιτικής και νομίζω ότι είναι σχετικό για τη δική σας επιτροπή λένε ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία με τα διάφορα δίκτυα και αναφέρουν ε, διάφορα δίκτυα που αναφέρα πριν ε, και τους φορείς εναλλακτικής απειλής διαφορών. Αλλά επίσης ε, αναφέρεται και πόσο σημαντικό είναι να προβάλλετε να προβάλλετε τα επιτέγματα του δικτύου. Επόμενη διαφάνεια. Υπάρχουν κάποιες άμεσες συστάσεις σε ό,τι αφορά το θέμα της προβολής Ανέφερα το Solvit, το Finet, μπορώ να φέρω και το Rapex που είναι ένα ακόμα δίκτυο Σάνκο, αλλά τα ECC ουσιαστικά δεν ε, αποτελούν ε, μια πολύ γνωστή ονομασία. Έτσι, λοιπόν, εντάξει, στα αγγλικά μπορεί να το γνωρίζουν κάποιοι, αλλά όχι στι άλλε γλώσσε, το ECC. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μια σύσταση να χρησιμοποιείται κάτι κοινό σε όλε τι γλώσσε. Και επίση, σύσταση λέει θα πρέπει να έχουμε εθνικέ τοσελίδε που θα είναι διαρθρωμένε με τον ίδιο τρόπο και θα μπορούν καταναλωτέ να αλλάξουν από τη μία χώρα στην άλλη και να βρίσκουν ακριβώ τι ίδιε πληροφορίε ε, στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, για να καταλάβουν ότι πρόκειται για δίκτυο και όχι μια λυσίδα απλώ μεμονωμένων κέντρων. Ε, προτείνεται επίσης ε, ένας ε, σχεδιασμός πρόθεσης ως ένα τμήμα του ετήσιου προγράμματος εργασίας και τονίζεται η σημασία της συνεργασίας με τους εμπορευμένους, με τις επιχειρήσεις πιστεύουν ότι υπάρχουν παράγοντες πολυπλησιασμού όπως παραδείγματος αεροδρόμια, τα λιμάνια, και διάφορες ταξιδιωτικά γραφεία κτλ και ε, πολλά σημεία συχνά ασκείται lobbying. Έτσι λοιπόν ε, τονίζουν πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με όλους αυτούς τους οργανισμούς. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε δύο ακόμη πτυχές. Αναφέρουν οι αξιολογητέ ε, το EDR, εναλλακτική επίλυση διαφορών, όπου θα πρέπει να έχουμε προαιρετική εξέλιξη. Γενικό Διευθυντή στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ εργάζεται για την ανάληψη ορισμένων νομικών πρωτοβουλειών στον τομέα αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν θα κάνουμε μία πρόταση, θα ληφθούν υπόψη συστάσεις. Και κάτι πολύ σημαντικό. Στο κάτω μέρος της διαφάνειας βλέπετε το θέμα των ε, Οφελών που προσφέρονται ε, από τα ΕΣΥ για ωφέλη για την κοινωνία. Εδώ πόσο κοστίζει η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, δηλαδή ε, αν έχουμε καταναλωτέ που προσπαθούν ε, να αγοράσουν διασυνοριακά. Πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν τίθεται το θέμα ότι και αυτή η πτυχή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όταν ε, λοιπόν εξετάζουμε ε, τα ωφέλη του δικτύου, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή, τα ωφέλη στην κοινωνία. Χαίρομαι που θα σα ενημερώσω ότι ήδη υπάρχουν ορισμένε ανεξελίξει δραστηριότητε. Υπάρχει μια εκστρατεία προβολή που ξεκίνησε αυτό το μήνα και ελπίζουμε να διαρκέσει όλο το καλοκαίρι, ίσως και περισσότερο. Σε 12 χώρες έχουμε θέσει εφαρμογή κάποια πιλωτικά προγράμματα, έχουμε και τυποποιημένες ιστοσελίδε και τις Κομισιόν αλλά και τις Εθνικές σελίδες και προσπαθούμε να δούμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στους καταναλωτές. Ήδη υπάρχει μια ομάδα μελέτης ε, μεταξύ του δικτύου CC και CPC δηλαδή όσων εκπροσωπούν ε, τους καταναλωτές και όσων θέτουν σε εφαρμογή την νομοθεσία και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα κράτη-μέλη. Στην επόμενη διαφάνεια αναφέρουμε το πρωτόκολλο ε, διαχείρισης των υποθέσεων, εσωτερικό έγγραφο αυτό, για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει streamlining των διαδικασιών και έχουμε παρομοιές διαδικασίες σε όλη την Ένωση. Και θέλω να αναφέρω επίσης ότι υπάρχει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν σκόπευε να είναι πιλωτικό πρόγραμμα εξ αρχής αλλά μετατρέπεται σε κάτι τέτοιο. Στην τελευταία σύνοδο του κατανοητές το 2010 είχαμε ένα εργαστήριο για θέματα ενοικίασης αυτοκινήτων. Ε, πολύ συχνά λαμβάνω καταγγελίες από σας και από τους σε τέτοια θέματα και εκ μέρους της Κομισιόν ε, τα εξετάζουμε και από ό,τι φαίνεται ο κλάδος αυτός για την ενοικίαση αυτοκινήτων ενισχύει πάρα πολύ ε, για την κακή φήμη. Έτσι λοιπόν ε, προσπαθούμε να έχουμε τώρα μία προσέγγιση φιλική προς το χρήστη και εξετάζουμε πώς μπορούμε να έχουμε εναλλακτική επίλυση διαφορών και πώς μπορούμε να παράχουμε πληροφορίες στους καταναλωτές ώστε να εκπροσωπούνται και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές ισότιμα. Στην τελευταία διαφάνεια βλέπετε το χρονοδιάγραμμα και τι συμβαίνει. Έχουμε μια διαβούλευση με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Ήδη ρωτήσαμε, ζητήσαμε από τις εσείς να συμμετέχουν στη μελέτη. Επευθύνθηκαμε στους διευθυντές της καταναλωτικής πολιτικής την περασμένη εβδομάδα στα κράτη-μέλη. Σήμερα είμαστε εδώ και φυσικά θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις από των διάφορων πορισμάτων. Θέλουμε να αναθεωρήσουμε τους στόχους στο δικτύου μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Και όπως το φθινόπωρο θέλουμε να το ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία και αν πάνε όλα καλά θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και θα έχουμε και συμφωνία με τα συγχρηματοδοτούτα κρατημέλη. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε τα επόμενα πέντε έτη να τα ξεκινήσουμε πιθανότατα με νέους στόχους και με μια αναθεωρημένη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Euh, σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ήταν πληρέστατη. Και καταδεικνύει πόσο πολυσύνθετο είναι το θέμα με το οποίο ασχολείστε. Θα ήθελα, εφόσον έχω το λόγο, να θέσω μία ερώτηση. Μιλήσατε πολύ για την ικανοποίηση των καταναλωτών, αλλά ταυτόχρονα για την έλλειψη κινήτρων για τις επιχειρήσεις ε, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα συνεργασίας με τις εθνικές και τις τοπικές αρχές. Οπότε, ρωτώ το εξής, ε, για τους προσεχείς μήνες, ε, τι προβλέπετε να γίνει και επίσης υπάρχουν θεμελιώδη προβλήματα όπως σε άλλους τομείς, τα οικονομικά προβλήματα. Είπατε ότι έχετε 30 φορές περισσότερες ανάγκες σε σχέση με αυτά που όντως γίνονται και αυτό καταδεικνύει ότι χρειάζονται ε, μεγαλύτερες προσπάθειες ε, για να ικανοποιηθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και θα μπορούσατε ίσως να αναπτύξετε περαιτέρω τις σχέσεις που έχετε με τις εθνικές αρχές. Μετά θα ακούσουμε και τη Μαργαρίτα που θα θέσει άλλη μια ερώτηση και θα σας δώσουμε τον λόγο. Ε, Ευχαριστούμε αυτά που μας είπατε και για τη μελέτη. Τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Ειδικά τα ζητήματα που αναφέρατε με απασχόλησαν και εμένα. Μήπως ε, με όλα αυτά τα δίκτυα μπερδεύονται οι καταναλωτές και μετά έχουμε και τις ενώσεις καταναλωτών. Θα γεμίσουμε οργανώσεις που ασχολούνται με τους καταναλωτές. Και δεν ξέρει κανείς σε ποιον θα απευθυνθεί τελικά. Το αναφέρατε. Είπατε επίσης πως θέλετε να βρείτε μια λύση. Ελπίζω να βρούμε και πρέπει να βρούμε επιγόντως λύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χρηματοδότηση. Νομίζω αν χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα λεφτά θα είναι καλύτερο από το να τα σκορπάμε σε διάφορα ανταγωνιστικά δίκτυα. Άλλο θέμα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Πώς θέλετε να την ε, ενσωματώσετε, γιατί πρέπει να συνδεθείτε και με αυτήν. Και θυμάμαι πριν από τέσσερα χρόνια νομίζω είχα πάει στην Ουάσιγκτον και συζήτησα εκεί πέρα με οργανώσεις καταναλωτών και εκεί πέρα είδατε, είδαμε τι γίνεται όταν έχει κανείς νομοθετικά εργαλεία όπως την ε, συλλογική προσφυγή. Τώρα οι συνάδελφοι που είναι μονίμως κατά λείπουν κιόλας από εδώ πέρα, αλλά βλέπετε πως ε, εκεί πέρα οι επιχειρήσεις προσπαθούν από μόνες τους να βρουν μια εναλλακτική λύση γιατί δεν θέλουν να μπλέξουν με ομαδικές προσφυγές και προτιμούν τις εναλλακτικέ. Είχαμε εδώ πέρα μια ιδεολογική διαφωνία για την οποία λυπούμε γιατί Βεβαίως θα πρέπει η συλλογική προσφυγή να αποτελεί τελευταία λύση, αλλά όταν υπάρχει συμπεριφέρονται διαφορετικά και οι επιχειρήσεις. Και νομίζω πως πρέπει να στηριχθούν όλα αυτά τα δίκτυα. Εμένα με εντυπωσίασε το πόσο ισχυρά είναι αυτά τα δίκτυα και πόσο χρηματοδοτούνται από τις επιχειρήσεις κτλ. Ευχαριστούμε, κυρία Χανσλίνγκ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον... Ε, ευχαριστούμε για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα ήθελα να θέσω διάφορες ερωτήσεις. Νομίζω ότι προκύπτουν διάφορα προβλήματα διότι δεν ε, υπάρχουν ε, δεν γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι υπάρχουν αυτά τα δίκτυα. Εγώ στη χώρα μου όταν ε, ρωτώ κάποιους αν γνωρίζουν την ύπαρξη του δικτύου, με κοιτάζουν εμβρόντιτοι, ούτε καν γνωρίζουν ότι υπάρχουν. Άρα η εκστρατεία ευαισθητοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία μα. Είπατε ότι στην Πολωνία έχει ξεκινήσει η εκστρατεία. Μα εγώ η ίδια προσπαθώ να βρω λεπτομέρειε για αυτή την προϊούσα εκστρατεία και δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βρω περισσότερες λεπτομέρειες, άρα υπάρχει επικοινωνιακό πρόβλημα. Οι καταναλωτές σίγουρα δεν ενημερώνονται επαρκώς. Ίσως οι ενώσεις καταναλωτών δεν ε, δραστηριοποιούνται ε, επαρκώς για την ενημέρωση των καταναλωτών το δίκτυο. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να τα χρησιμοποιούν. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ρίξουμε το βάρος σε αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης να δραστηριοθούμε περισσότερο. Ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε και ένα δίκτυο όπως το Solvit και το Rapex, ε, να έχουμε δηλαδή το ίδιο όνομα για τα δίκτυα σε όλες τις χώρες. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές ως προς την ονοματολογία των δικτύων. Πάλι για να ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές. Κατόπιν μας είπατε ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι πάντοτε πρόθυμες ε, δεν ε, απαντούν σε επιστολές ε, καταγγελιών για επανόρθωση. Μου φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του εναλλακτικού μηχανισμού διευθέτησης διαφορών και θεωρούν ότι είναι χρονοβόρα και περίπλοκη η δικαστική διαδικασία. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του μηχανισμού εναλλακτική διευθέτησης των διαφορών, ούτως ώστε να μην να παραμένουν ευυπόλοιπτες ενώπιον του δικαστηρίου ε, και να χρησιμοποιούν ε, τον εναλλακτικό αυτό μηχανισμό. Προτείνω λοιπόν να οργανώνονται συχνότερα αυτές οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Γνωρίζω ότι οικονομικός πώς είναι προβληματική αυτή η ιδέα, αλλά για να έχουμε καλά αποτελέσματα και ικανοποιημένους καταναλωτές θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Αυτό που μόλις μας είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, με την άποψή σας. Μήπως είναι αυτό μια ωραία πρόκληση για την Πολωνική Προεδρία. Θα υποφεληθούμε από το ότι είσαστε, θα αναλάβετε την Προεδρία. Απάντηση. Ναι, ναι, δίκιο έχετε. Θα να διαβιβάσω το μήνυμα στην Πολωνική Προεδρία και είμαι πεπισμένη ότι θα το εξετάσουμε σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Πρόεδρος. Το είπα αυτό διότι συχνά στη Γαλλία λέω ότι περιμένουμε πολλά από την Πολωνική Προεδρία και το πολωνικό λαό για να αλλάξει η θεώρηση των πραγμάτων που είχαμε και έχουμε ακόμη στη Γαλλία. Θα συνεργαστούμε λοιπόν και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και προς κεκλημένους μας. Ποιος είναι τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι. Ωραία, θα ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Μανχώτε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας ε, και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων για τα διάφορα ζητήματα που σχολίασα στην παρουσίασή μου. Προσπάθησα να συλλέξω όλα τα ερωτήματα. Αν παραλείψω κάτι, να μου το επενθυμίσετε. Παρακαλώ. Πρώτον, σχετικά με το ε, στάδιο στο οποίο βρίσκονται αυτά τα δικτύα των καταναλωτών. Δεν πρόκειται για ενώσεις καταναλωτών. Δύο τρίτα των κέντρων διαχειρίζονται από εθνικές αρχές, από υπουργεία θέλετε. Μόνο το ένα τρίτο βρίσκεται σε επίπεδο ένωση καταναλωτών. Το δίκτυο της Πολωνία, Παραδείγματο χάρη το διαχειρίζεται μια εθνική αρχή στη Γερμανία. Ε, ε, είναι διαφορετικά τα πράγματα διότι υπάρχει μια ανεξάρτητη οργάνωση που διαχειρίζεται και το γαλλικό και το γερμανικό δίκτυο. Συστεγάζονται, αν θέλετε, αυτά τα δίκτυα και χρησιμοποιούν τι ίδιε υποδομέ. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ δομέ για τα δίκτυα. Πλην δεν υπάρχει ανταγωνισμό σε αυτό το τομέα. Δεν γνωρίζω να υπάρχει καμία ένωση καταναλωτών που να ασχολείται με διασυνοριακά καταναλωτικά ζητήματα. Δεν ανταγωνίζονται τι εθνικέ Ένωσε Καταναλωτών, δηλαδή αυτά τα δίκτυα. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει καμία διένεξη ως προς τη χρηματοδότησή τους. Τα κράτη-μέλη επιλέγουν ε, ποια είναι η καλύτερη οργάνωση αμφιτρίων και ε, είμαστε πεπισμένοι ότι γίνεται καλή κατανομή από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Όταν μιλάμε για τα θέματα εμπιστοσύνη. Γιατί δεν χρησιμοποιούν τον εναλλακτικό μηχανισμό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα έλεγα ότι πρόκειται μάλλον για θέμα νοοτροπίας. Στις σκανδιναβικές χώρες 80% των διαφορών λήγουν σε επίπεδο εναλλακτικού μηχανισμού διευθέτησης διαφορών. Δεν πηγαίνουν καν στα δικαστήρια, διότι και οι επιχειρήσει και οι ιδιώτες επιθυμούν να ε, κλείσουν μια συμφωνία. Ε, αν δούμε τώρα τις αντιλήψεις σε κάποιες άλλες ε, νότιες κυρίως χώρες, ε, θα διαπιστώσουμε ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, η απόφαση που ενδεχομένως θα ληφθεί και θα εφαρμοστεί δεν θεωρούν ότι μπορεί να προκύψει μέσω μιας φιλικής διευθέτησης διαφορών και γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τον εναλλακτικό μηχανισμό. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγή νοοτροπίας. Τώρα, αν θα πρέπει να καταστήσουμε υποχρεωτική και δεσμευτική την απόφαση που λαμβάνεται από τον ε, εναλλακτικό μηχανισμό διευθέτηση διαφορών, αυτό είναι στα παρέμβαση στην Εθνική Ενόμη Τάξη. Δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικέ ε, οι αποφάσει, γιατί έχουμε τα δικαστήρια, έχουμε τι εθνικέ ε, διαδικασίε διαχείριση των καταγγελιών, διευθέτηση των διαφορών. Θα πρέπει να έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, λοιπόν, οι αποφάσει του εναλλακτικού μηχανισμού. Για τι συλλογικέ αγωγέ, αναφερθήκατε σε αυτό. Λειτουργεί ω το σύστημα στη ΣΥΠΑ, βέβαια υπάρχει και διάσταση απόψεων. Ε, ναι, ναι, λειτουργεί καλά, αλλά υπάρχει και μία πίεση ε, που οδηγεί σε αύξηση της χρήσης του ελεκτικού μηχανισμού διευθέτησης διαφορών. Έτσι δεν είναι. Απάντηση. Το ε, ε, έχουμε επίγνωση αυτού. Ε, Μία άλλη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής άρχισε να εξετάζει αυτό το θέμα και ε, σε πάνω από τα μισά κράτη-μέλη υπάρχουν εναλλακτικοί μηχανισμοί διευθέτησης διαφορών και το θέμα μας τώρα είναι με ποιο τρόπο μπορούμε με συστηματικό τρόπο να παράσχουμε λύσεις, όχι μόνο για, τις, για τους καταναλωτές ή για θέματα καταναλωτών, αλλά και για θέματα ανταγωνισμού η ήδη υπηρεσιακά η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή εκπονεί μια ενιαία προσέγγιση, μια δέσμη κανόνων που θα εφαρμόζονται και στους δύο τομείς και με το που περατώσουμε αυτές τις εργασίες ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα βήματα στον τομέα αυτό. Για τη χρηματοδότηση. Είναι όντω ένα θέμα η χρηματοδότηση και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης. Βεβαίως είναι ζωφερό το οικονομικό κλίμα ε, και θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά με τα ορόσημα που σας παρουσίασα σήμερα, ε, μάλλον τα δεδομένα που σας παρουσίασα σήμερα, ελπίζω να πείσω εσάς και όλους όσους λαμβάνουν αποφάσεις στο Συμβούλιο ε, να λάβουν τις αποφάσεις που επιθυμούμε για τη χρηματοδότηση. Επίσης, θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά με επιπρόσθετα κονδύλια. Ε, λένε ότι ε, υπάρχει υπερσυμφόρηση στα κέντρα, ότι δεν μπορούν να χειριστούν άλλε υποθέσει αυτά τα κέντρα και άρα ε, όλοι προχωρούν προσεκτικά με αυτέ τι εκστρατείε ενημέρωση. δηλαδή, αν διαφημίσουμε τι υπηρεσίε μα, θα έχουμε περισσότερε καταγγελίε από του κατάλληλε, όμω δεν μπορούμε να τι διαχειριστούμε στη συνέχεια, γιατί δεν έχουμε επαρκή στελέχωση. Οπότε δεν είναι το ζήτημα μόνο σε επίπεδο διαφήμιση και ενημέρωση και προφανέστατα αυτό συνεπάγει το μεγαλύτερο κόστο, ε, αλλά είναι θέμα πόρων. Ε, μέχρι ε, πόσες μάλλον καταγγελίες μπορούμε να διαχειριστούμε μέσα σε αυτά τα κέντρα. Ε, σας ευχαριστούμε εξάλλου και για την υποστήριξη της ιδέας σχετικά με το ενιαίο όνομα του, για όλα τα δίκτυα και ελπίζουμε ότι θα στεφτεί με επιτυχία αυτή η ε, εκστρατεία. Για 12 χώρες έχουμε 200.000 ευρώ μόνο, είναι ελάχιστη η πόρη. Τώρα, αυτά που, σε σχέση με αυτά τα κονδύλια που χρησιμοποιεί το Google παραδείγματο χάρη, ε, δεν είναι τίποτα. Αυτή η έβρεση που προβλέπεται σε διάφορες γλώσσες στο Google για την υποβολή καταγγελιών. Ε, όλα αυτά συνεπάγονται επενδύσεις ε, και ελπί, ε, έχουμε και πληρωμένες διαφημίσεις στο διαδίκτυο και ελπίζουμε ότι μέσα στο Google θα αρχίσουν να εμφανίζονται όλο και περισσότερο εικονίδια αυτών των δικτύων στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης για να γίνουν και δοκιμές από τους καταναλωτές. Αν αποδείξουν την αξία τους τα δίκτυα θα έχουμε καλά αποτελέσματα και ψημένη χρήση από τους καταναλωτές. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Σε παρακαλώ να μου θυμίσετε, αν τυχόν παρέλειψα κάτι, να μου το πείτε. Με Ευχαριστώ πολύ. Μας μένει λίγος χρόνος ακόμη. Σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε για τα χρήματα 200 εκατομμύρια ευρώ για 12 χώρες. Πραγματικά μοιάζει πρόκληση, δηλαδή αν θέλετε να εργαστείτε Τελάμε τόσο λίγα μέσα. Είναι δύσκολο, αλλά είναι δυνατό. Ε, το περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο ψήφισε το σχετικό προπολογισμό. Μπορείτε να βασίζεστε λοιπόν στο Κοινοβούλιο και θα είμαστε στο πλευρό σα. Και φυσικά πάντα σα υποστηρίζει και η δική μα Επιτροπή. Και καθώ ε, έδωσα τη σκητάλη και στην Πολωνική Προεδρία θα έχουμε ίσω και κάποια μέλη του Συμβουλίου μαζί μα. Αυτό θα είναι καλό για τη χρηματοδότηση και για το ευρωπαϊκό όραμα. Μήπως ε, κάποιοι από του ευρωβουλευτές θέλουν να θέσουν κάποια άλλη ερώτηση, όχι. Μάλιστα, θα κλείσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε. Καλή τύχη και καλό κουράγιο και θα τα ξαναπούμε σύντομα γιατί πράγματι αυτή η πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω όχι μόνο πρέπει να έχουμε τους υλικούς αλλά και τους ανθρώπινους πόρους στη διαθήκη και πρέπει να συνεργαζόμαστε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα πολύ συντονισμένα για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ε, υπάρχουν πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ παρόντα, αλλά θα ήθελα να πω ότι σήμερα το απόγευμα στις 3 έχουμε δει συνεδρίαση των εισηγητών και των σχεδόν εισηγητών για την ε, έκθεση για την προστασία των καταναλωτών και κλεισμένο το θυρών, έκθεση ΒΑΜΠ ε, και στις στις 3.30 θα συνεχίσουμε τις δημόσιες ε, εργασίες μας ε, για την ε, έκθεση του κυρίου Κρότσμαν. Και έχουμε και την ακρόαση στις 4. Γεια σας.